Το θέμα στην εμερήσια διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Μπέλετ για τη σταθερότητα της αγοράς και το αποθεματικό στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Κύριε Μπέλετ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Καλό απόγευμα. Νομίζω ότι σήμερα Όλοι έχουμε το βλέμμα στραμμένο ε, στην ελληνική κρίση και αυτό ίσως ε, επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς όμως δεν περιμένει αλλαγή του κλίματος ε, και θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στον αγώνα μας κατά των αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε λοιπόν να εισαγάγουμε ένα ε, σύστημα αυτόματης διόρθωσης με αυτό το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Είναι ένα σημαντικό βήμα για αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας εκπομπών το οποίο μετά την οικονομική κρίση ή λόγω της οικονομικής κρίσης ε, σχεδόν ε, κατέρευσε. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν νέα κίνητρα για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στη μείωση των εκπομπών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ε, για να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας και το στόχο να έχουμε μείωση κατά 30% των εκπομπών μέχρι το 2030. Θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι για να έχουμε και μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση ε, στη διάσκεψη των Παρισίων στα τέλη του έτους. Με το πρώτο αυτό βήμα ενισχύεται πράγματι σημαντικά η θέση μας. Η μεταρρύθμιση αυτή την οποία θέλουμε να εγκρίνουμε συνεπάγεται ότι θα έχουμε μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική που θα συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η μετάβαση ε, σε παραγωγή με χαμηλές εκπομπές άνθρακα σημαίνει ε, περισσότερες επενδύσεις. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό εκτός ένωσης ε, που δεν, από εταιρείε που δεν χρειάζεται να αγοράσουν δικαιώματα ε, εκπομπών. Άρα υπάρχει εδώ πραγματικά κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει μεν ανάπτυξη αλλά και ανταγωνισμός. Υπάρχουν σημαντικές παρεκκλήσεις και σημαντικές νέες πρωτοβουλίες που συμφωνήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ε, μάλλον στο πλαίσιο αυτής της ε, πρότασης, έχουμε ε, κάποιες παρεκκλήσεις για και θα σας πω τρεις αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα παρέκκληση ελεύθερα δικαιώματα για τομέα της υπαρχής ισχύω. Δεύτερον, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, 2 δις ευρώ. Είναι ένα ταμείο που δημιουργείται τώρα για περαιτέρω επενδύσεις σε συγκεκριμένα κράτη που έχουν ε, χαμηλότερο ε, από το μέσο όρο του ΑΕΠ και επίσης ε, επένδυση, κατανομή με, στις χώρες αυτές που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Επομένως, αν όλα πάνε κατευχήν, την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Κανιέτε, ο αρμόδιος επίτροπος, ε, θα καταθέσει μια νέα πρόταση και συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου, παρέχοντας εγγυήσεις ε, κατά της διαρροής άνθρακα. Και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά των θερμοκηπιακών αερίων. Είναι καλή πρόταση, ισορροπημένη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Κανιέτε τους υπολείπους ε, συνεργάτες του από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, της οποίας ηγείται να ευχαριστήσω και τη Λετωνική Προεδρία ε, και τους πρέσβεις γιατί πολύ επαγγελματικά χειρίστηκαν το όλο ζήτημα. Να ευχαριστήσω τους κύριους Γκεμπράν και Χάουτ, Γκέπχαρτ, Εύη, Κάλλονεν και όλους τους άλλους Λαβία, τον πρώτο τη Επιτροπή Ένβη, συγητή είτε τον Κιωταγιάννη. Εξαιρετική ήταν η συνεργασία με όλου αυτού, γιατί δεν θα είχαμε καταφέρει χωρί αυτού να έχουμε αυτή την έκθεση σήμερα. Ευχαριστώ και τώρα ο Επίτροπος για την κλιματική δράση και την ενέργεια, κύριε Επίτροπε Κανιέτε. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, για μένα είναι ικανοποίηση που είμαι και πάλι ενώπιόν σας στα πλαίσια τη συζήτηση για το αποθεματικό σταθερότητα της αγοράς. Εφόσον το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με αυτά που επιτέχθησαν στο Συμβούλιο, θα αποτελέσει το απόθεμα αυτό τμήμα του συστήματος εμπορίας ε, εκπομπών. Θα είναι λοιπόν ακρογωνίος λίθος του συστήματος, διότι τα τελευταία χρόνια οι διακυμένοι στην αγορά δεν επέτρεψαν στο σύστημα αυτό να έχει το αναγκαίο αποτέλεσμα για να γίνουν οι επαρκείς επενδύσεις σε χαμηλού άνθρακα τεχνολογίες. Αυτό το στόχο προσπαθεί να επιτύχει, αυτό το πρόβλημα να επιλύσει περισσότερη ευελιξία αυτή η πρόταση, ούτως ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς στο σύστημα. Και τα επόμενα χρόνια οι τιμές να έχουν την κατάλληλη κατεύθυνση για να επιτύχουμε τους στόχους μας, να μειωθούν μακροπρόθεσμα οι εκπομπές. Αυτό το αποθεματικό θα μας ε, εξασφαλίσει να μην χάνουμε ευκαιρίες για να έχουμε μείωση των εκπομπών. Ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές για την εργασία τους, ιδιαίτερα ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Μπέλετ και τους συνεργάτες του και τον κύριο Ταγιάννη και τους κοιόδης των πολιτικών ομάδων για τις προσπάθειές τους. Ο συμβασμός των οποίων καταλήξαμε είναι μια ρωμαλαία λύση με βάση σημαντικά στοιχεία για να επιτύχουμε τη σταθερότητα της αγοράς. Να σας πω ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλεγε ότι το 2021 θα άρχισε να λειτουργεί αυτό το αποθεματικό. Κατά την συζήτηση πολλοί βουλευτέ ζήτησαν να υπάρξει νωρίτερα λειτουργία και αποφασίσαμε το 19 να αρχίσει να λειτουργεί. Επίσης, αυτά τα οποία θα αφαιρεθούν από την αγορά, τα δικαιώματα που θα αφαιρεθούν θα πάνε σε αυτό το αποθεματικό. Αυτά λοιπόν τα 900 εκατομμύρια που αποσύρθηκαν από την αγορά μεταξύ 14 και 16 δεν θα πάνε στην αγορά το 2020 όπως προέβλεπε αρχικά η πρόταση. Τα δικαιώματα που δεν θα έχουν χορηγηθεί θα πάνε επίση στο αποθηματικό. Άρα θα μειωθεί ο κίνδυνο πτητικότητα στο σύστημα. Η σημασία τη καινοτομία για μένα είναι ένα από τα πιο ουσιώδη στοιχεία αυτή τη συμφωνία. Επίση αναφέρεται στο κείμενο. Στο πλαίσιο θεώρηση του συστήματο εμπορία των εκπομπών θα δούμε εάν τα 50 εκατομμύρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα αξιοποιηθούν για να ενθαρρύνουμε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Στο κείμενο επίσης αναφέρουμε τη σημασία που έχει η ανταγωνιστικότητα και ο κίνδυνος που σημαίνει διαρροή άνθρακα για τον κλάδο. Τα δύο στοιχεία αυτά σας διαβεβαιώ ότι είναι σημαντικά και θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια της πρώτας ανθεώρησης του συστήματος ETS. Όλα τα στοιχεία που ανέφερα θα επιτρέψουν μια καλή δομή για αυτό το αποθεματικό και θα ενισχύσουν το ETS στο μέλλον. Επιτύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο με αυτό το συμβασμό που μας επιτρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στην ανθεώρηση του συστήματος ETS για την περίοδο 2030. Πέρυσι δεσμεύτηκα ενώπιόν σας να βάλω τα σημεία του πανέργειας που σχετίζονται με το ETS σε μια συγκεκριμένη πρόταση όσο ταχύτερα ε, επιτευχθεί συμφωνία για αυτό το αποθεματικό. Και είναι πρόθεσή μου τον Ιούλιο λοιπόν να υποβάλω πρόταση με βάση την συνένεση που επέτυχαν αρχικά των κυβερνήσεων τον περασμένο Οκτώβριο. Η πρόταση αυτή θα είναι σημαντικό τμήμα της εργασίας που πρέπει να εκτελέσουμε για να έχουμε μια ενεργειακή πολιτική συνδεδεμένη με την πολιτική κλίματος. Αυτά είναι προτεραιότητες για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, ο κύριος Σταγιάννη, για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπέλετ, για την εξαιρετική του δουλειά, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία και να ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την δουλειά του και τη συνεργασία του, διότι με την τελική αυτή συμφωνία καταλήξαμε σε ισορροπία μεταξύ της πολιτικής για το περιβάλλον και της πολιτικής για τη βιομηχανία. Έχουμε προβλέψει σημαντικά μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν να αποφύγουμε το επιπλέον κόστο για τι επιχειρήσει, αυτά που θα προκύψουν από την επιβολή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το κλίμα. Να θυμίσω όλο ιδιαίτερω τι διατάξει για τη διαρροή του άνθρακα και το Ταμείο για την Καινοτομία που θα πρικοδοτηθεί με 50 εκατομμύρια για την ε, ανταλλαγή δικαιωμάτων, ε, ανταλλαγή αερίου του θερμοκηπίου. Για την κλιματική μας πολιτική πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία μεταξύ δύο πτυχών. Για το μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει ο αριθμός των ε, όσων θα προβλέψουμε για τι ανακυκλώσιμες πηγές ενέργεια και την αντιστάθμιση τη τιμή για το διεξίδιο του άνθρακα. Ελπίζω ότι θα, πρέπει να, θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την βιομηχανία μα προστατεύοντά την από τη μετατόπιση επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης. Και για τα έμεσα κόστη θα πρέπει να βρούμε ε, ένα εναρμονισμένο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ κρατών με αρνητικέ συνέπειε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ελπίζω, ολοκληρώνοντα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτέ τι προτάσει της μεταρρύθμισης του συστήματος ε, με το στόχο 40% μείωση των αερίων του θερμοκοπίου μέχρι το 2030. Πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι υπάρχει κι άλλος ένας στόχος γενικός για το 20% της μεταποιητικής βιομηχανίας έως το 2020. Χωρίς βιομηχανία δεν υπάρχει δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λίζα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Μπέλετ αλλά και τον Τζοβάνι Λαβία πρόεδρο της Επιτροπής και τον εισηγητή της Ήτρε Αντώνιο Ταγιάννη και ευχαριστώ και όλους τους άλλους που συμμετείχαν. Το ΕΛΚ φυσικά θα υπερψηφίσει αύριο το κείμενο αυτό. Είναι καλή πρόταση της Επιτρόπου Χέντεγκάρντ και με τη βοήθεια του κυρίου Αρία Κανιέτε που τη διαδέχθηκε βελτιώθηκε η πρόταση. Η πρόταση είναι φιλόδοξη. Πιο φιλόδοξη από την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένοι την επικρίνουν λέγοντας ότι δεν πάει αρκετά μακριά. Αλλά κοιτάξτε, ξεκινάμε δύο χρόνια νωρίτερα. Και επίσης ε, διαφορετικά από ότι προέβλεπε αρχική πρόταση τα δικαιώματα που βγαίνουν από την κυκλοφορία θα μπουν στο αποθεματικό και δεν θα κατανεμηθούν μέχρι το 2020. Και όσα δεν κατανεμηθούν μέχρι το 2020 και αυτά θα μπουν στο αποθεματικό. Αυτό νομίζω ότι είναι φιλόδοξη διαδικασία για να προστατεύσουμε το κλίμα, για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα ETS. Ε από την άλλη πλευρά, και συμφωνώ, κάναμε διευκρινήσεις που βοηθάνε να αποφύγουμε τη διαρροή άνθρακα. Δεν θέλουμε οι ενεργοβόρες ε, βιομηχανίε να μετακατασταθούν. Θέλουμε μέσω καινοτομία, μέσω των νεωτέρων τεχνολογιών και γι' αυτό έχουμε τα benchmark και γι' αυτό θα χρησιμεύσει και το ταμείο που επέβαλε το Κοινοβούλιο παρά πολύ έντονε αντιδράσει. Εμεί ω Κοινοβούλιο θέλουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο σε αυτή τη δυσχερή οδό και παρακαλώ να δεχθεί αυτή μας την προσφορά, αυτό το απλωμένο χέρι ο κλάδος και να μην ε, απορρίψει αυτή μας την πρωτοβουλία. Α, αυτή είναι η οδός που οποία πρέπει να βαδίσουμε και ελπίζουμε η Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα, γιατί είμαι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να προστατεύσει, να κάνει φιλόδοξε προσπάθειε προστασία του κλίματο, αλλά να δώσει τη δυνατότητα και στον κλάδο να συνεχίσει να λειτουργεί. Έτσι θα αποτελέσουμε πολύ καλό παράδειγμα και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λίκη Πρόεδρε. Ο κύριο Γκρότε, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ Ήβο, ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο έδρασε με υπεύθυνο τρόπο για αυτό το σημαντικό θέμα, διότι το ETS θα βοηθηθεί από αυτό το αποθεματικό. Και η ομάδα μου ενωμένα θα το στηρίξει το επαθηματικό λοιπόν αυτό επιτέλους θα επιτρέψει να αναπνεύσει το ETS. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι συγκυριακές ε, διακυμάνσεις. Γιατί ε, προηγουμένως το σύστημα αυτό βαζόταν σε ε, κρατική λειτουργία. Αυτό ήταν μια δομική αδυναμία. Το διορθώσαμε τώρα με αυτό το επαθηματικό και είναι πολύ καλό που 1,5 δικαιώματα θα πάνε στο αποθεματικό, θα βγουν από την αγορά. Άρα θα αντιμετωπίσουμε τη δυσχέρεια αυτή. Νομίζω πως είναι ρεαλιστική αυτή η πολιτική για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις τεχνολογίες που θα μειώσουν τις εκπομπές και πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές πλαίσιο για όσους θέλουν να επενδύσουν. Οπότε ήταν καιρός να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και δίνουμε και ένα σαφές μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο και προς την COP21 ότι χρειαζόμαστε μια καλή βιομηχανική πολιτική όπως την είπα στα Γιάννη Αποτιμία και προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ότι αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Ότι αυτά δεν αλληλοαποκλείονται. Είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένο και επαναλαμβάνω δράσαμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο και το επιτύχαμε. Η ομάδα μου, όπως ήδη αναφέρθηκε, συμφωνεί με το συμβιβασμό για την ανακτήρια ε, ημερομηνία αυτού του ε, αποθεματικού και συνολικά μπορούμε νομίζω να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική προχωράνε. Και περιμένω την πρότασή σας ε, κύριε Επίτροπε Κανιέντε, ελπίζω πριν το καλοκαίρι, Ίσως μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ρώτησα τον κύριο Σεύκοβιτ, Σε συνεδρία της Επιτροπής είπε ναι, ναι, ναι, πριν τις διακοπές. Το ρώτησα, ναι, αλλά ποιας χρονιά στις διακοπές. Μου είπε φέτος και ελπίζω ε, να είναι φέτος, όντως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Παρακαλώ να παραμένετε στον χρόνο αγόρευσή σας. Ο κύριος Ντάνκαν για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το σύστημα ανταλλαγή ήταν μια από τι εμβληματικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είχε καθόλου άνεμο στα πανιά του. Έτσι λοιπόν να πω στον κύριο Μπέλετ ότι είναι δύσκολο να μεταρρυθμίσουμε ε, ένα ε, δυσλειτουργικό ε, πολιτικό σύστημα, ένα δυσλειτουργικό σύστημα, μια επιλογή πολιτικής, αλλά οι προτάσεις του ούτως ή άλλως δεν θα βελτιώσουν ε, θα βελτιώσουν εν μέρη με την συμβολή των πολιτικών ομάδων ε, όσα προτείνονται. Το 2019 νομίζω είναι μια καλή ε, αφετηρία και με τα εκατομμύρια που προτάθηκαν νομίζω καλώς κινηθήκαμε. Η διαδικασία αυτή δεν θα λειτουργούσε με αυτά τα ποσά. Επίσης, το, η νέα φάση του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών θα θέσει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για τη λειτουργικότητα του ε, ε, του συστήματος αυτού. Εάν θέλουμε να επιτύχει τα αποτελέσματά του και να δημιουργηθούν παρόμοια συστήματα και στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, εάν σφάλουμε, αν επιβάλλουμε, επιβάλλουμε υπερβολικό άχθος σε αυτούς που περισσότερο εκπέμπουν, θα έχουμε πάλι προβλήματα. Χαίρομαι που υπάρχουν λοιπόν όροι σε σχέση με την διαρροή του άνθρακα και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κάνουμε σωστές επιλογές. Δεν θέλουμε να έχουμε απλώς περιορισμό των εκπομπών αποκλείοντας βιομηχανικούς κλάδους που είναι τόσο σημαντικοί για πολλά μέρη της Ένωσης. Με όλα αυτά πρέπει να πω ότι είμαστε στη σωστή πορεία. Θα πρέπει τουλάχιστον να επιτύχουμε εξωσημείωτη πρόοδο, εάν θέλουμε να ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών και ειδικά πριν φτάσουμε στη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι. Γι' αυτό ανυπομονώ για την ψηφοφορία αύριο και πρέπει να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό σε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Ένα βήμα προόδου που είναι απλώς το πρώτο. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θα ε, έρθουν μπροστά μας και στα Σύνοδο του Παρισιού. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά ο κύριο Φέρα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλετ, τον ε, πρόεδρο Λαβία και τον συνάδελφο κύριο Μπράντι για την εξαιρετική δουλειά τους ε, για το έγγραφο αυτό το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, ε, δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του συστήματο αυτό που είναι σημαντικό με την εκχώρηση αδειών, χωρί όμω η αγορά να στρεβλώνεται και να υπάρχει η απεριόριστη, το απεριόριστο δικαίωμα για τις εκπομπές. Για οικονομικούς λοιπόν σκοπούς η αλλαγή του συστήματος είναι σημαντική γιατί με τις διαπραγματεύσεις που είχαμε σε σχέση με αυτή την νομοθετική πρόταση είδαμε να δημιουργηθεί ένα σταθερότερο και πιο προβλέψιμο πλαίσιο με περιβαλλοντικούς στόχους και λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτομίες των πράσινων τεχνολογιών. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσουν πριν από το 2020 να προτείνουν ένα ταμείο καινοτομία για να προωθηθεί η έρευνα και νέε τεχνολογίες με χαμηλή καταναλώση άνθρακα. Πρέπει να προετοιμάσουμε από σήμερα τις αυριανέ τεχνολογίες. Και αυτό φαίνεται ότι και η σταθεροποίηση του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών θα αρχίσει να λειτουργεί νωρίτερα από ό,τι είχε ανακοινώσει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020, δηλαδή το 2019. Σας συγχαίρουμε γι' αυτό και πραγματικά θα πρέπει αμέσως στο παθηματικό για τη σταθεροποίηση της αγοράς να ε, προβλεφθούν 900 εκατομμύρια ε, δικαιώματα τα οποία προβλέφθηκαν για να, για να αντιμετωπίσουν την πίεση της αγοράς. Αύριο καλούμαστε να εγκρίνουμε αυτή την νομοθετική πρόταση και να αποστείλουμε μια ένδειξη στους εξωτερικούς μας εταίρους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρά και υπεύθυνα το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Κύριε Επίτροπε, να μην ξεχνάμε την κατεπίγουσα ανάγκη να έχουμε μια ε, παγκόσμια συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές που να είναι δεσμευτική και να προβλέπει στόχους χώρα. Θα πρέπει, Επίτροπε, να μην ξεχνάμε ότι δεν ε, έχουμε ε, ότι είναι δική μας ευθύνη μάλλον εμείς οι Ευρωπαίοι να ξεκινήσουμε αυτή την διαδικασία. Δείξατε την πλήρη προθυμία σας και αφοσίωσή σας προς αυτό το στόχο και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον Σάφα Φερέιρα. Παρακαλώ, έχετε 30 δευτερόλεπτα κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο. Είπατε ότι η αγορά για τι ανταλλαγέ δικαιωμάτων είναι βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Εγώ έχω να, αντιμετω... να αναφέρω σωρό παραδείγματα που η αγορά αυτή λειτουργήσε για τον αντίστροφο σκοπό, για να δοθούν περισσότερα δικαιώματα εκπομπών. Μα λέτε λοιπόν σε ποια περίοδο συγκεκριμένα το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών συγκεκριμένα ενίσχυσε την, ε, το στόχο αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου, εάν αποτύχει αυτός ο μηχανισμός, τι μπορείτε να προτείνετε ως λεκτικό εργαλείο. Ευχαριστούμε κύριε φρέια για 30 λεπτά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Η θέση της ακροαριστεράς είναι αντίθετη με το μηχανισμό αυτό, το σύστημα. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό επιτρέπει πραγματικά να μειωθούν οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου και να αντιμετωπιστούν οι κλιματικέ αλλαγέ. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να ε, ε, μπορέσει να γίνει πραγματικότητα χάρη σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό η κυρία Κούλωναν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Βέβαια, Πρέπει να πω ότι τελώ υπό κάποια σύγχυση. Έχουμε ε, κάποιους ε, στόχους ε, μη φιλόδοξους, έχουμε οικονομική ύφεση, ήταν ε, άτολμο το σύστημα εμπορίας. Το σύστημα δεν λειτουργήσε και τώρα προσπαθούμε να το τροποποιήσουμε μπορεί και να μην είναι η ιδανική λύση, είναι όμως ένα πιθανό βήμα ε, προς τα εμπρός. Είμαι ε, πραγματίστρια και αισιόδοξη και γι' αυτό σκέφτομαι να ψηφίσω υπέρ της πρότασης. Στη δική μου πολιτική ομάδα γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές ε, που δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ούτε μετά από τις διορθώσεις ε, και ευελίξτεμα, ότι θεωρώ ότι δεν θα είναι. Σας ευχαριστούμε και τώρα για 1,5 λεπτό. με κύριο Σέικχαουτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλετ για την εξαιρετική του δουλειά. Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να πετύχει κανεί συμβαστική πρόταση για το σύστημα ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων. Είναι μια συζήτηση που όλου μα κοιτάζει στην Ολομέλεια, αλλά και αλλού. Και τελικά συνήθω δεν καταλήγουμε σε συμβαστική λύση. Αυτή τη φορά καταφέρατε να πετύχετε ένα συμβασμό και νομίζω ότι πραγματικά σα αξίζουν συγχαρητήρια. Σα ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε εμεί ω πράσινοι. Μπορούμε να στηρίξουμε την συμβαστική αυτή πρόταση. Θα υπερψηφίσουμε λοιπόν γιατί θεωρούμε ότι είναι βελτίωση αυτό που είχαμε προηγουμένω. Ε, Όμω η δουλειά μα μόλι ξεκινάει. Διότι ξέρουμε ότι έχουμε ένα μηχανισμό για την σταθερότητα τώρα, αλλά είναι τεράστιο το πλεόνασμα των αδειών που ε, κρέμονται άχρηστε ε, και παραμένουν ε, πάνω από την αγορά σε ένα σύννεφο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ε, λύσει την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πρότασή τη. Διότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνήθω για το σύστημα αυτό αργούν, αλλά α δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και μια ερώτηση προ τον κύριο Κανιέτα, τον Επίτροπο πραγματικά διαβάζουμε ειδήσει ότι λίγο πολύ μεταβάλλεται μια από τις προτάσεις σας που ήταν αρκετά πετυχημένη ως τώρα. Δηλαδή τις ε, άδειε που δεν έχουν ε, αποδοθεί ακόμη, δεν έχουν δοθεί σε κάποιον να πάνε κατευθείαν στο αποθυμητικό. Στην ίδια διαδικασία λέτε ότι θέλετε 250 εκατομμύρια από τις άδειε για ένα νέο μέρο του αποθυματικού. Δηλαδή ήδη μειώνεται η φιλοδοξία μας για τους στόχους το 2020. Ε, έχω καταλάβει λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε. Διότι καταλάβαμε ότι την επόμενη εβδομάδα ήδη η γενική μας αίσθηση θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές προτάσεις. Δηλαδή ότι το πλεόνασμα των αδειών που δεν χρησιμοποιούνται θα πάνε απευθείας στο αποθυματικό. Ελπίζουμε να ακολουθήσετε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε κυρία Εύη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί, το σύστημα ανταλλαγή ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Ένα παράλογο σύστημα που μέσω τη αγορά επιτρέπει να, δεν επιτρέπει να υλοποιηθούν σοβαρές και υπεύθυνε πολιτικές για το κλίμα. Δεν έχουν θαρρυνθεί οι επιχειρήσεις να ε, επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες και έχει και παράπλευρες συνέπειες που είναι καταστροφικές πρώτα απ' όλα την ε, κερδοσκοπία. Η αγορά των δικαιωμάτων βρίσκεται στα χέρια brokers που εκμεταλλεύονται και τον τομέα του περιβάλλοντος. Πέρα από τις απάτες που ευνοεί και την φοροδιαφυγή και έχει προκαλέσει 5 δις ευρώ απόλυση στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, η έκθεση που εκπονήθηκε πρόσφατα για το σύστημα αυτό δείχνει πόσε παράνομε ε, δράσει υπάρχουν σε σχέση με το σύστημα αυτό, ακριβώ γιατί είναι άλλη η φύση των ε, τίτλων. Είναι ανήθικο λοιπόν οι στόχοι που ορίζονται ω βιώσιμοι και προσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών που αφορά το σύστημα αυτό. Ακόμη και ο Πάπα ζήτησε να ε, δώσουμε περισσότερη σημασία στην ανθρώπινη διάσταση του προβλήματο και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε μόνο με την οικονομική συνιστόσα. Ευχαριστούμε κυρία Ντορνανό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να δείξει ότι δεσμεύεται να σεβαστεί τις προτάσεις και τις συστάσεις του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Δημιουργώντας μία αγορά ETS. Ο μηχανισμός αυτός έπρεπε να επιτρέψει μία σταδιακή αύξηση της τιμής του άνθρακα και έτσι να αποσβέσει να χρηματοδοτήσει την μεταρρύθμιση της οικονομίας μας, αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι τιμές κατέρευσαν. Η δημιουργία ενός αποθεματικού είναι μόνο ε, συμπτωματική και επιφανειακή θεραπεία. Η πραγματική συζήτηση θα έπρεπε να αφορά τις ποσοστώσεις και το πώς ρυθμίζουμε τις εκπομπές. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν ήδη κάνει μεγάλη προσπάθεια ενώ οι αναπτυσσόμενε χώρε μολύνουν όλο και περισσότερο. Και σύντομα θα φτάσουν στο επίπεδο εκπομπών των χωρών του Βορρά. Το σύστημα του κιότο είναι λατωματικό και οι βιομηχανίε μα και η ανταγωνιστικότητά μας υποφέρουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μπαλώματα τεχνοκρατών. Ευχαριστώ, λέει ο Α, βλέπω μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Από τον κύριο Φερέιρα. Όχι, Φαρία. Φαρία. Δέχεστε μια μπλε κάρτα παρακαλώ. Α, ωραία, ευχαριστώ. Τρία δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς την ε, κυρία συνάδελφο. Μα δεν βλέπετε ότι αυτό που κάνουμε με το MSR είναι να βοηθήσουμε να λειτουργήσει το σύστημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Ξέρουμε ότι δεν πάει καλά. Άρα πρέπει να το διορθώσουμε και να συγκρίνουμε για παράδειγμα τι γίνεται στη χώρα σας σε σχέση με τη χαλιβουργία της ε, Σουηδίας. Η δική μας βιομηχανία είναι και καθαρότερη και αποτελεσματική και πιο ανταγωνιστική. Και πέρα από το ETS και τώρα το MSR έχουμε και ένα πολύ υψηλό φόρο διοξιδίου του άνθρακα. Δεν βλέπετε όλα αυτά ωφελούν όταν κάνεις το σωστό. Κυρία μου, 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε, λέει η Πρόεδρος. Μα πώς να υπερασπιστούμε ένα σύστημα όπου αυτοί που μολύνουν περισσότερο είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και δεν έχουν δεσμευτικού στόχους. Αυτό βαραίνει στο δικό μας κλάδο. Είμαστε λοιπόν σε μειονεκτική θέση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αποθωτικοί από οικονομική άποψη αλλά ρεαλιστέ από περιβαλλοντική. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Μπάλσο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το ETS, ε ο αρχικός στόχος ήταν να είμαστε αποτελεσματικοί και να επιτύχουμε τους στόχους μας το 2020. Έχουμε μια συνολική ποσόστοση και οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα είναι υπερβολικά φιλόδοξη. Όμως η Ευρώπη είναι υπεύθυνη μόνο για 19% των εκπομπών στον κόσμο. Άρα τι σημασία έχει τι θα τηρήσουμε εμείς. Οι λίγες επιχειρήσεις μας που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα καινοτόμε, δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και κλείνουν. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν άνεργοι και μετά εισάγουμε χάλβα από την Ινδία. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να απευθυνθώ και στην Υπουργό, γιατί έδωσα όθηση για να πετύχουμε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι στην αίθουσα αυτή πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπέλετ και όλου του συντονιστέ των πολιτικών ομάδων, αλλά και την Προεδρία, του, την εργασόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, γιατί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή συμφωνία σε αυτό το θέμα. άκουσα στη συζήτηση αυτή κάποιοι να επικρίνουν το σύστημα ΙΤΕΣ, το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Ξέραμε ότι δεν ήταν τέλειο, ξέραμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση, αλλά αυτή είναι πραγματική μεταρρύθμιση του συστήματο. Ε, το αποτελεσματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, επιτρέπει η ε, εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα να παραμένουν σε επίπεδα που να είναι αποδεκτά και να δώσουν και ένα κίνητρο στο βιομηχανικό σύστημα ώστε βιώσιμα να επιδιώξει την μείωση των εκπομπών. Σήμερα μιλάμε για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και ελπίζουμε ότι αύριο θα εγκριθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες αυτής της Ολομέλειας. Ένα όμως είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό Τότε το συζητάμε την παραμονή τη αναθεώρησή του. Ε, ο Επίτροπο έχει αναλάβει μια δέσμευση και είμαστε βέβαιοι ότι θα την τηρήσατε. Όμω πρέπει πάνω απ' όλα πριν από την διάσκεψη των μερών 21 στο Παρίσι να φροντίσουμε να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ευρώπη να παραμείνει πρωταγωνίστρια στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και με ε, το εργαλείο αυτό που θα εγκρίνουμε αύριο να επιβεβαιώσει την ισχυρή της βούληση να υπάρχει η βιωσιμότητα για το βιομηχανικό μας σύστημα και στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακρογωνίω λίθος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το 45% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιοριστεί. Όμως το σημερινό σύστημα έχει πολλά ε, ελαττώματα, όπω φάνηκε από τον άδειε που παρέμειναν αδιάπτε στην αγορά, ενώ ε, συνεχίζει να υπάρχει η ίδια, το ίδιο επίπεδο εκπομπή αερίων. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να μεταρρυθμιστεί και να γίνει ένα μηχανισμό ελέγχου των εκπομπών αλλά και προώθηση των επενδύσεων στι καθαρέ τεχνολογίε όπω τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και προβλεψιμότητα για το σύστημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πετύχουμε του στόχου μα για τι κλιματικέ αλλαγέ. Αλλά ταυτόχρονα να παράσχουμε και περισσότερη σταθερότητα στην αγορά και την βιομηχανία. Πιστεύω ότι το αποθεματικό για τη σταθερότητα τη αγορά είναι το κατάλληλο εργαλείο για να πετύχουμε τη σταθερότητα τη αγορά. Αυτή ήταν η θέση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γι' αυτό στηρίξαμε την εισαγωγή του όσο το δυνατόν συντομότερα, ε, μεταφέροντα τα δικαιώματα για τι εκπομπέ δεξιδίων του Άθρακα ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα και ε, τι άδειε όταν δεν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση. Θα πρέπει να είναι και πιο ευέλικτο και πιο σταθερό το σύστημά μα, ώστε να πετύχουμε του στόχου μα για το κλίμα. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα με τη σωστή ισορροπία που να επιτρέπει στι βιομηχανίε και τι εταιρείε να δρουν ε, σωστά με μια βιώσιμη πράσινη οικονομία στην Ευρώπη που να αποτελέσει μοντέλο και πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι να δείξουμε στους πολίτες και τις βιομηχανίες μας και τις μελλοντικέ γενιές στον δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα. Τον κύριο Ουβιεντόφσκι. Ναι. 30 δευτερόλεπτα κύριε μου. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα το οποίο μόλις ακούσαμε. Γιατί θα πρέπει να είναι όσο το τον υψηλότερε οι χρεώσει για τι εκπομπέ. Υπάρχουν κάποιε χώρε που η οικονομία του στηρίζεται στον άνθρακα και αν αυτή είναι η άποψή σας, πώς ε, πιστεύετε ότι μπορεί να αντισταθμιστεί η παραδοσιακή οικονομία άνθρακα. Τι είδους αλληλεγγύη μπορεί να μένει κανείς από εσάς. 30 ε, δευτερόλεπτα για την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ τη βορειοδυτική Αγγλία και θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι ήταν πολύ σημαντικά τα ορυχεία στην ε, περιφέρειά μας όπως και οι τεχνολογίες και η βιομηχανία. Εμείς θέλουμε όλους αυτούς τους κλάδους να τους προστατεύσουμε με τον εξυγχρονισμό ETS και το MSR και προβήκαμε σε δράση με το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Θα έχουμε και το μηχανισμό σταθερότητας μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη, ώστε και το κλίμα να προστατεύσουμε και τις ανανεώσιμες ενέργειες να προωθήσουμε και τους βιομηχανικούς κλάδους να προστατεύσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Κυρία Βυσνιεύσκα τώρα έχει το λόγο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι κατά αυτού του αποθεματικού και την σταθερότητα της αγοράς. Είναι κάτι το οποίο βασίστηκε σε λάθος νομική βάση πολύ απλά. Θα έπρεπε να υπόκειται στην ε, ομοφωνία εντός του Συμβουλίου. Θα είναι πολύ αρνητικό για τη χώρα μου. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία έχουν υψηλά, ε, υψηλές ανάτομο. Αυτό το αποθεματικό θα χτυπήσει σκληρά τους Πολωνούς λόγω της συγκεκριμένη ενεργειακής μας δομής. Και αυτό σημαίνει ότι το κόστος θα είναι άκρος δυσανάλογο σε σχέση με τα κέρδη. Επίσης, αντιτίθεμε σε αυτού του είδους τους τεχνητούς ελέγχους τιμών. Τα δικαιώματα εκπομπών είναι φθηνά λόγω της οικονομικής κρίσης και για κανέναν άλλο λόγο. Δέχεστε, λέει η Πρόεδρο. Ο κύριος Τσάνι, ε, ερώτηση με για κάρτα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα αυτά που υπόθηκαν. Και τώρα θέλω να με εξηγήσετε. Γιατί είμαστε κατά να θεωρούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί. Γιατί δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση. Δεν επιδιώκουμε να βαδίσουμε μια διαφορετική οδό. Με συγχωρείτε 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε. Με βάση την συνθήκη κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να αποφασίζει το ενεργειακό του μείγμα. Στην Πολωνία ε, ο κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του και ο εξορρυκτικός κλάδος και ε, ο ενεργειακός. Τα προτινόμενα μέτρα θα αυξήσουν τη διαφορά μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων κρατών μελών. Ευχαριστώ, ο κύριος Φέντερ, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ. Καταρχάς, Ευχαριστώ τον κύριο Κερ συγγνώμη, να εκφράσω ευχαριστήσεις του κυρίου Γκερμπράντι, αλλά και τι δικές μου. Ο κύριος Γκερμπράντι δεν είναι, μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπέλετ γιατί κατέληξε σε έναν ε, καλό συμβασμό. Καλό και ε, ρωμαλαίο συμβασμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει περισσότερα. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό ο συμβασμό γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε ότι καταραίει εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Όμω, ορισμένοι συνάδελφοι λένε ότι διώχνουμε τι επιχειρήσει μα από την Ευρώπη. Όμω έχουμε ακόμη τέτοιε επιχειρήσει στην Ευρώπη και αυτέ είναι αυτέ που έκαναν ήδη τι μεταρρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι η Κίνα τα πάει καλύτερα για τη Χαλιβουργία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Συγγνώμη, όχι, συγγνώμη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι καλύτερε ε, για το χάλιβα και η Κίνα είναι καλύτερη για το τσιμέντο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έχουμε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βιομηχανία. Ευχαριστώ, Λε Ένα λεπτό, η κυρία Κανέτσουνα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την πρόταση αυτή. Σκοπός της είναι να αλλάξει τη δομή του ETS, του συστήματος ανταλλαγής δικαιωμάτων, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πλεόνασμα διών που έχει δημιουργηθεί από το 2009. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το στραβό σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών διορθώνεται. Ε, βεβαίως, Έχω ακόμη πολλούς ενδιασμούς, διότι το ETS μπορεί να είναι απλώς ε, μία προσωρινή λύση. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς στόχους και συγκεκριμένους ε, για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν έχουμε ακόμη αρκετά μέτρα για τη διαρροή του άθρακα. Χρειάζεται ε, μια πολιτική συμφωνία για το ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο. Αν δεν συμφωνήσει και η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλοι μεγάλοι ρηπαίνοντες στον πλανήτη για δεσμευτικού στόχους, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε μόνοι μας με το ευρωπαϊκό σύστημα. Χρειάζεται μια παγκόσμια λύση. Ευχαριστούμε κύριο Έριξον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι και εγώ συχνά αμφέβαλα για το σύστημα αυτό επανειλημμένος. Το σύστημα αυτό που έχουμε στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό. Ένα σύστημα που αφορά διαφορετικά κρατημέλη όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι από πολύ καιρό δυσλειτουργεί. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια σωστή αποτίμηση και να δούμε ποιες ε, είναι, ποια είναι τα λογικά συμπεράσματα. Χαίρομαι για τη δουλειά που έγινε στην Αρμόδια Επιτροπή από τους και εισηγητές. Τώρα έχουμε μια ένα πραγματικό βήμα προόδου, μια, ε, ένα τρόπο να κάνουμε κάποια διαφορά στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει και νομίζω να ε, υλοποιήσει όσα θα συμφωνηθούν. Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε αδράνεια, πρέπει να περάσουμε σε δράση. Θέλουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί με πρόσθετα μέτρα όπως προτείνονται και ελπίζουμε ο κύριος Κανιέτα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ε, κάποιες ιδέες πολύ σύντομα ώστε να δείξουν ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες της σε αυτό το τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω γαλάζια κάρτα ζητήθηκε, αλλά συνάδελφος ήδη είχε μιλήσει, οπότε θα δώσω το λόγο για να λεπτό στην κυρία Ρίντ. Ε, κυρία Πρόεδρε, στηρίζει ε, ο εισηγητής ε, την πρόταση της Κομισιόν για ένα αποθεματικό σταθερότητα της αγοράς, θεωρώντα ότι οι διακοιμάσει στην αγορά έτσι θα ρυθμιστούν και θα έχουμε μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα και σταθερότητα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Αυτό είναι αναλυθέ. Μηχανισμοί όπως το ETS, τα, τα όπιστο βαρύ δικαιώματα και το MSR είναι από τα βασικά αίτια της φτωχοποίησης των βιομηχανιών μας. Η ιδέα ότι αυτό το σύστημα εμπορίας θα στείλει μηνύματα στις αγορές και θα προωθήσει την ε, διατήρηση της ενέργειας και ε, τεχνολογίες ε, χαμηλής, χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν έχουν πετύχει και συνεχίζει να αποτυγχάνει αυτό το σύστημα. Παρ' όλα αυτά προτείνει τώρα η Κομισιόν αυτό το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται όμως είναι ότι ένας μηχανισμός αγοράς απαιτεί ρυθμίσεις ρυθμιστικέ παρεμβάσει για τη διατήρηση των επιπέδων των τιμών και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονό ότι θα πρέπει αυτόνομα να ορίζουν τι τιμές οι αγορέ. Δεν θα πρέπει να στηρίξουμε κλεισίματα λουκέτα επιχειρήσεων. Θα πρέπει ε, την ε, φθήνουσα οικονομία να την αναζωογονήσουμε με μια τελείω διαφορετική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ακούστε συνάδελφοι, λόγω τη πίεση χρόνου όταν ζητείτε μπλε κάρτα θα δίνω το λόγο μόνο σε όσου συναδέλφου δεν έχουν ήδη μιλήσει. Κυρία Κέρλινγκ, νομίζω ότι μιλάτε αργότερα. Επομένως δεν θα σας δώσω τώρα τη δυνατότητα να εκφραστείτε με μπλε κάρτα. Επόμενος ομιλητής ε, Στούγκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μαγνήτης ε, ε, ατυχιών Έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες, έχουμε δημοσιονομική κρίση, τώρα έχουμε και το ETS που ποτέ δεν λειτουργήσε, ούτε λειτουργεί, ούτε θα λειτουργήσει. Αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι Κινέζοι ή άλλοι, από άλλες υπήρους πάντως. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνουμε τόσο ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια που οι επιβάτες ε, προτιμούν άλλε αεροπορικές εταιρείε που έχουν πιο φθηνά εισιτήρια. Το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ πραγματικά υποφέρει λόγω αυτής της κατάστασης. Στις Βρυξέλλες πολλοί λένε απλά λόγια αντί να κάνουν πράξεις και με τη θεωρία του άνθρακα αν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να γίνει με τους τεχνοκράτες και γραφειοκράτες που θα πρέπει να τους διαρρεύσουμε κάπου αλλού. Θέλετε να απαντήσετε σε μπλε κάρτα παρακαλώ, λέει πρόεδρος. Κύριε Στούγκερ, με ακούτε. Δέχεστε μπλε κάρτα. Δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Φρουντζουλίτσα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Είπε κάτι ο κύριος Στούγκερ. ότι αυτό το πλεόνασμα δικαιωμάτων οδήγησε το σύστημα σε αποσταθεροποίηση. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του αποθεματικού της σταθερότητα της αγοράς θα σταθεροποιήσει την αγορά τελικά. Απάντηση. Ακούστε, το μόνο που λέω εγώ είναι ότι ένα θα είναι το αποτέλεσμα, η αποσταθεροποίηση. Και αυτό το βλέπουμε με το ελληνικό ζήτημα, το ζήτημα της μετανάστευσης. Όλα αυτά αποσταθεροποιούν την κατάσταση. Και οι δράσεις της Ένωσης σε όλους αυτούς τους ε, τομείς αποτυγχάνουν. Και το ίδιο θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει να το καταλάβει αυτό κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπέλετ, που κατέληξε σε αυτή τη συμφωνία με όσους τον βοήθησαν για τη δημιουργία αυτού του επαθεματικού σταθεροποίησης της αγοράς. Θα μπορούν έτσι οι εταιρείε να επενδύσουν στις τεχνολογικές λύσεις χαμηλής καταναλώσης άνθρακα, παραμένοντας βέβαια υψηλά ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει σήμερα να ακούσουμε τις ανησυχίες του βιομηχανικού κλάδου που εκτίθεται στους κινδύνους της διαρροής του άνθρακα. Θα πρέπει κύριε Επιτροπέ αυτό το πολύ σοβαρό στοιχείο να το ε, παρακολουθήσετε. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αναθεώρηση της οδηγίας του συστήματος που θα προτείνεται ήδη την επόμενη εβδομάδα. Θέλω και να εκφράσω μια συγκεκριμένη ανησυχία. Ήδη πολλέ εταιρείε έχουν καταβάλει τεράστιε προσπάθειε, έχουν μειώσει κατά το ίμιση τι ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα τα τελευταία χρόνια και ξέρουν ότι δεν μπορούν πλέον να πάνε παραπέρα. Δεν έχουν την απαραίτητη τεχνολογία, έχουν κάνει ήδη τι ε, απαραίτητε προσπάθειε. Το να τι υποχρεώσετε να είναι ακόμη πιο φιλόδοξε σημαίνει ότι θα τι βάλετε σε πολύ μεγάλε δυσκολίε. Ιδίω σκέφτομαι την χαλιβουργία. Ε, στην ομάδα μα το ΕΛΚ θέλουμε και ένα ταμείο καινοτομία με τους ε, με πληστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα κάνει να δημιουργήσει ένα τέτοιο ταμείο με 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ακόμα πολύ αδύναμο, αλλά ήδη είναι μια πρικοδότηση. Το ταμείο αυτό, εφόσον αρχίσει να υπάρχει, τουλάχιστον θα μπορέσει να στηρίξει τις μελλοντικές τεχνολογικές λύσει. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδης. Ως μητέρα ενός ε, αγοριού θα ήθελα ο γιος μου να μεγαλώσει σε ένα καθαρό περιβάλλον και να έχει δυνατότητα να βρει ποιοτική απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτή είναι η ισορροπία που πρέπει να επιτύχουμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχο του ETS. Όταν πριν από 10 χρόνια το δημιουργήσαμε, ως το πιο σημαντικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι τώρα δεν θα είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ναι μεν επιτύχαμε μείωση των εκπομπών, αν και ίσως αυτό να οφείλεται στην οικονομική κρίση, αλλά από την άλλη μεριά το ETS ε δεν κατάφερε να στείλει επαρκή μηνύματα για την κατεύθυνση των τιμών για να υπάρξουν καθαρές επενδύσεις. Άρα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και έχουμε ένα τεράστιο πλεονάσμα δικαιωμάτων. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε το MSR τάχιστα. Το αργότερο το 2019 θα έλεγα. Αυτό το MSR θα πρέπει να δώσει ακριβώς σταθερότητα. Να αποφευθεί η διακύμανση των τιμών. Να στείλει δηλαδή ισχυρό μήνυμα στην αγορά, να βοηθήσει τον κλάδο να προγραμματίσει τις επενδύσεις του, σε καινοτόμε και καθαρέ τεχνολογίες. Η επιτυχία ή η αποτυχία του ETS θα επηρεάσει τα επίπεδα εκπομπών και τελικά την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν το σύστημα να είναι αποτελεσματικό για να μειώσουμε όντως τις εκπομπέ με αποδοτικό τρόπο και να παραμείνουν ανταγωνιστικέ επιχειρήσεις μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γκέρλινγκ. Το ETS δεν είναι τέλειο βέβαια, αλλά είναι το βασικό μέσο πολιτικής που έχουμε ως Ένωση και είναι ενδιαφέρον ότι όλοι όσοι το επικρίνουν απλώς το επικρίνουν δεν προτείνουν εναλλακτικέ. πώς αλλιώς θα μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου άρα καταλήγω ότι δεν ανησυχούν δεν ενδιαφέρονται για να μειωθούν τα αέρια αυτά σε πολλές περιπτώσεις το γνωρίζω γιατί λένε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα αέρια θερμοκηπίου αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό ότι ακόμη και σήμερα λέγονται αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχει καμία σχέση με το πώς πιστεύουν ότι έχουν τα πράγματα οι περισσότεροι επιστήμονες. Ένα θέμα να αναφέρω. Διαρροή άνθρακα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα της ανταγωνιστικότητας βιομηχανίας μας. Και δεν είναι ασύμβατο με τους στόχους κλιματικής αλλαγής. Και είναι πραγματικά ενοχλητικό να υπάρχει αυτή η διάσταση επιχειρημάτων. Πρέπει να περάσουμε σε χαμηλού άνθρακα τεχνολογίες. Μας το είπε ο κύριος Τίμερμανς. Πρέπει να έχουμε ευφυεί πράσινε τεχνολογίε. Χθες τα είπε. Αλλά γι' αυτό πρέπει να γίνουν επενδύσει, πρέπει να είναι κερδοφόρε επιχειρήσεις και πρέπει να έχουμε και τις αναγκαίε πιστώσει. Ευχαριστώ λέει πρόεδρο. Πρόεδρος. Ένα λεπτό. Η κυρία Έρνστ Ευχαριστώ πολύ. Είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Όπως το βλέπουμε. Το βασικό είναι όμως να είμαστε αισιόδοξοι. Να πούμε ναι, είναι μισογεμάτο. Καλό που κάτι γίνεται και που κάτι θα γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Καλό είναι που θα αρχίσει το σύστημα νωρίτερα, κατά δύο χρόνια νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν έτσι έναν ευέλικτο μηχανισμό. Αυτό είναι πρόοδος. Και τα οπισθοβαρή δικαιώματα του θα μπουν στο αποθεματικό. Και αυτό είναι καλό. Και χρειάστηκε πολλής αγώνας για να το επιτύχουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον υπερβολικό κίνδυνο στο αποθεματικό. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουν γίνει περισσότερα γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν ασυνέπειες με αυτόν τον τρόπο στο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να υπάρξει αύξηση της τιμής για να έχει αποτελεσματικότητα το σύστημα. Να έχει επιπτώσεις. Και η εμπορία δικαιωμάτων, το εμπόριο δικαιωμάτων να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή. Ούτως ώστε τελικά το ποτήρι να γεμίσει μέχρι πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλμερ ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει κρίση ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Λόγω της υψηλής τιμής της ενέργειας. Κλείνουν επιχειρήσεις, ανεργία και οι επενδύσεις πάνε εκτός Ευρώπης εντελώς. Και παρόλα αυτά κύριε Πρόεδρε, εμείς εδώ μέσα σήμερα συζητάμε πολιτικές που έχει σαφή στόχο να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την τιμή της ενέργειας. Εμείς θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα μειώσουμε την τιμή της ενέργειας. Φαίνεται συνάδελφοι ότι έχουμε διάθεση να αυτοκτονήσουμε οικονομικά όπως είπε ο συνάδελφος μου, Dr. Reed οποιοδήποτε λεγόμενος μηχανισμός αγοράς που ξεκινάει με ένα εκ των προτέρων καθορισμένο επίπεδο τιμών και που χρειάζεται διαρκής παρεμβάση για να επιτύχει αυτή την τιμή δεν είναι μηχανισμός αγοράς. Είναι ένα εξαιρετικά ε, ε, βαρύ και ακριβό σύστημα φορολογίας του άνθρακα. Ας έχουμε λοιπόν είτε ένα ξεκάθαρο φόρο στον άνθρακα ή καθόλου φόρο στον άνθρακα. Ευχαριστώ κύριο Μπέι. Ένα λεπτό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ, δεν λειτουργεί. Κύριε Μπέι. Κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφε, το σύστημα ανταλλαγής ε, δικαιωμάτων εκπομπών δεν λειτουργεί. Ε, Όμω αντί να το καταστρέψει, οι τεχνοκράτε μαζί με τον κύριο Σούλτ προτίμησαν να δημιουργήσουν ένα αποθεματικό για τη σταθερότητα αγορά για να αντιμετωπίσουν αυτή τη λειτουργία. Αυτή η αυτορύθμιση της αγοράς που τόσο πολύ αρέσει στους ευρωκράτες τελικά κατάληξε να είναι μια ομολογία αποτυχίας Για τις βιομηχανίε μα αυτή η λύση φαίνεται να συμπιναμεί με έμεσο φόρο και έμεση φορολόγηση. Όμως ε, αυτό το σύστημα βλάπτει ε, του, εμάς και όχι τους ανταγωνιστές μας εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν τα οικολογικά προσχήματα για τη μείωση των εκπομπών ε, διοξείδου του άνθρακα να ε, παραδεχτούμε ότι γίνονται ένα αντικείμενο εμπορίας όπως οποιοδήποτε άλλο οι απαταιώνες αυτοί με το στρεβλωμένο αυτό σύστημα επιτρέπουν να γίνει μια τεράστια απάτη με πάνω από 5 δις βρω κέρδος για τους ε, Αβί Μπεν Έζρα και τον Ψηρή Λαστρίκ λόγου χάρη. Οι φωνές του λαϊκού μετόπου δεν εμπόδισαν την έκθεση Ταγιάννη αυτή στην Επιτροπή Ήτρε δυστυχώς. Το ίδιο και η έκθεση Μπέλετ. Γκριζίμπ. Συζητούμε τη μείωση των εκπομπών για πάρα πάρα πολύ καιρό. Το ETS ε, κάποια επιτυχία είχε, μείωσε κάπως τις εκπομπές, αλλά γνωρίζουμε ότι έχει πέσει η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών λόγω της οικονομικής κρίσης. Χρειάζονται λιγότερα δικαιώματα. Ήμουν αντίθετος ε, αρχικά σε αυτό το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς επειδή πιστεύω ότι διαστρεβλώνει την ασφάλεια δικαίου. Το MSR ε, γνωρίζαμε ότι σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021, όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Φθινοπονίου Συμβουλίου για το κλίμα. Διάσκεψη κορυφής για το κλίμα. Υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε, παραλαμβάνω αυτό το αποθεματικό να λειτουργεί από το 2021. Επίσης, Υπάρχει και μια απόφαση για τα βαρύ δικαιώματα, τα οποία πλέον μπαίνουν σε αυτό το αποθεματικό. Και αυτό όμως διαστρεβλώνει την ασφάλεια δικαίου. Ανησυχεί πολλοί κόσμος και για τη διαρροή άνθρακα. Την ε, κατάσταση επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο Παρίσι, αν και ελπίζουμε να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία. Δεν θα πρέπει όμως να αλλάζουμε συνεχώς τα συστήματα έτσι όπως μας έρχεται κάθε φορά. Πρόεδρος, δεν βλέπω την κυρία Γκαρθία Πέρεθ, άρα θα περάσω στον επόμενο μιλητή για ένα λεπτό, ο κύριος Τόσενόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε η συζήτηση τι μέλη γενέστε με την εμπορία εκπομπών, ε, δικαιωμάτων εκπομπών δεν είναι ένα νέο ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι κάπως δύσπιστος απέναντι στο κατά πόσον αυτό το αποθεωματικό θα βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος ε, εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, διότι δεν νομίζω ότι καθοδηγητά από την αγορά και δεν είναι και βιώσιμο μακροπρόθεσμα αυτό το σύστημα. Δεν μου αρέσουν ε, ούτε ε, ε, οι παρεμβάσεις αυτές που μπορούν, πιστεύω, να διαταράξουν την οικονομία εν γέννη. Συμφωνώ για τις, τα δωρεάν αυτά δικαιώματα και την πρόταση του εισηγητή. Και πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή την αρμόδια φάνηκε ότι πρέπει να αλλάξει άρδινο ο κανονισμός για το ETS. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρος κύριο Κάρινς για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Επίτροπε Συνάδελφοι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση και ε, εμπορικών εταίρων και τώρα είμαστε και σε διαπραγματεύσεις με έναν ακόμη μεγάλο εταίρο, τις ΗΠΑ. Βασική προϋπόθεση της αμερικανικής πολιτικής είναι να ρίχνουν τις τιμές. Ενώ η ενεργειακή στόχη για μας είναι να έχουμε στο δυνατόν χαμηλότερες εκπομπές ε, αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι όμως αυξάνουμε τις τιμές της ενέργειας. Αυτό δυσχεραίνει πολύ τη ζωή των βιομηχανιών μας. Πώς να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ όταν έχουν χαμηλότερες τιμές εκεί. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία, το αποδεικνύει και η επιστήμη για την ανθρωπότητα. Είναι σημαντικό να μειωθούν τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα για να αντιμετωπιστούν παράλληλα και οι κλιματικές αλλαγές. Εμείς όμως οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και για την ανταγωνιστικότητα των, του μηχανικού μας κλάδου. Έτσι λοιπόν, πιέζοντα να μειωθούν οι εκπομπέ, ε, τελικά μπορεί να πιέζουμε προ τα πάνω τις τιμέ τη ενέργεια, κάνοντα την ε, τον τομέα της ενέργειας να είναι μη ανταγωνιστικό. Μπορεί να χρειάζονται εξαιρέσει ή παρεκκλήσει εκεί, ώστε να μην εξάγουμε προϊόντα και αρχίσουμε να εισάγουμε βιομηχανία. Δεν είναι αυτό ο στόχος μας, φαντάζομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Παολούτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μακρά οικονομική κρίση έχει αποδυναμώσει και προκαλέσει κρίση στο σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών. Ο τιμό των ποσοστώσεων και τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα έχει πέσει πάρα πολύ. Η τιμή αυτή, η χαμηλή τιμή, δεν δίνει κίνητρα για μελέτη τη καινοτομία και για ανανέωση και για βιώσιμε λύσει. Γι' αυτό το επαθεματικό για τη σταθερότητα τη αγορά δίνει την εξασφάλιση τη βιομηχανία ότι μπορεί να υπάρχει σταθερά και προβλήματα 50 εκατομμύρια ποσοστώσεις για τις ε, βιομηχανικές λύσεις τι καινοτόμε λύσει που θα προβλέπουν χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Αυτό είναι καλό και για του περιβαλλοντικού μα σκοπού, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και για το μηχανικό μέλλον τη Ευρώπη. Το απαθηματικό τη σταθερότητα τη αγορά βέβαια είναι ένα πρώτο μέτρο, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει αμέσω να μεταρρυθμιστεί συνολικά το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών. Ακούμε την υπόσχεση που εκφράσατε, Επίτροπε, να περάσετε πριν από τη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι σε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Ζούρμπου, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Κιώδης για την εργασία τους για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε κάτι που να ικανοποιεί όλα τα κράτη-μέλη γιατί υπάρχουν διαφορές στις οικονομίες μας. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βασικών μας ε, βιομηχανιών. Είναι λοιπόν πολύ ουσιώδης αυτές οι διαφορές. Στη χώρα μου υπάρχει σημαντική έκθεση στις υψηλές τιμές άνθρακα και επιπτώσεις από αυτό. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αν μπορούμε να δώσουμε κάποια οικονομική στήριξη, κάποιες αντισταθμίσεις στους κλάδους που φύγονται από αυτό το έμεσο κόστος του ETS. Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό όταν θα αναθεωρηθεί ο μηχανισμός αυτός. Ο μηχανισμός είναι πολύ σημαντικός για την Ένωση στην ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία προσέγγισης, ε, προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου. Θα δώσω το λόγο σε πέντε συναδέλφου. Πρώτο είναι ο συνάδελφο ε, Σον Κέλλη. Ένα λεπτό, κύριε Κέλλη, παρακαλώ. Πολύ σημαντική πρόταση και οπωσδήποτε θα πρέπει να συγχαρούμε ιδιαίτερα τον συνάλφο Μπέλετ. Τον είδα πώ εργάζεται και είναι πολύ λογικέ οι λύσει του που πρότεινε και θα βοηθήσουν τον Επίτροπο Κανιέτο να κάνει την έκθεσή του στις 15 Ιουλίου. Οπωσδήποτε οι στόχοι μα είναι δύο. Να μειώσουμε τι τις ε, εκπομπέ στην Ένωση κατά 40% μέχρι το 2030 και ο άλλο στόχο είναι να αναπτυχθεί κατά 20% του ΑΕΠ ε, ο κλάδος. Η βιομηχανία γενικά. Μπορούμε να τα επιτύχουμε και τα δύο αυτά. Δεν είναι παράλογα. Με βάση τις νέες τεχνολογίες και με βάση τις προτάσεις που έχουμε εδώ για το ETS και ιδιαίτερα για την ανακτήρια ημερομηνία που νομίζω ότι είναι πολύ καλή 2019. Μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Είμαι εισηγητή για την Ήτρε, για την κλιματική αλλαγή, για το Παρίσι και ελπίζω αυτό να βοηθήσει να επιτύχει συνάντηση αυτή κορυφή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ζουλ Παρνιό, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι συζητήσετε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την COP21, καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε Κανιέτη, και να επικροτήσω την δημιουργία του αποθεματικού για τη σταθερότητα τη αγορά άνθρακα που αύριο θα επικυρώσουμε με την ψήφα μα στην Ολομέλεια. Έτσι θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε το πλεόνασμα των δικαιωμάτων και να αποκαταστήσουμε σταδιακά την εμπιστοσύνη στον Ευρωπαϊκό Αυτό Μηχανισμό. Όμω, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, την COP21 στο Παρίσι και ήδη από τώρα γρήγορα γρήγορα θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή στην αγορά άνθρακα και να καθοριστούν ποσοτικοποιημένοι στόχοι μείωση ε, των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Με αυτό το εργαλείο, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ε, αποκαταστήσουμε τη διεθνή μας αξιοπιστία στον αγώνα μας κατά της αλλαγής του κλίματος. Αυτό είναι μια καλή προοπτική ε, εν ώψη του Δεκεμβρίου και της COP21. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η νομοθετική πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών προτείνει τη θέσπιση ενός αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς του συστήματος και ως λύση στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπών. οι εν λόγω ανισορροπίες οδήγησαν σε πλεόνασμα περίπου δύο δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών στην περίοδο εμπορίας δύο 2013-2020 και μειώνουν έτσι τα κίνητρα για επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα ο στόχος λοιπόν είναι να διορθωθούν οι ελλείψεις του συστήματος ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. η δημιουργία ενός αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το υπάρχον σύστημα θα φανεί όμως αναποτελεσματική εάν δεν προγραμματιστούν και χρηματοδοτηθούν σοβαρές και βιώσιμες επενδύσεις για εναλλακτικές πηγές ενέργειας. χωρίς τις παραπάνω επενδύσεις η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση της ευρωπαϊκής ένωσης σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα παραμείνει κενό γράμμα. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστούμε Γιάκοφτιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ψηφίσουμε την πρόταση αυτή θα θέλαμε να δούμε γρήγορα και την πρόταση της Επιτροπής, γιατί αυτό θα είναι το κατάλληλο βήμα προκειμένου να πετύχουμε τη σταθερότητα της αγοράς που επιθυμούμε. Η αντίφαση μεταξύ των αρχών για την μείωση των εκπομπών από τη μία και την ανάπτυξη της οικονομίας από την άλλη μπορεί να επιληθεί με επενδύσεις στην κοινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή τι θα κάνετε με τις επενδύσεις που έχουμε μπροστά μας και θα οδηγήσουν σε περισσότερη κατανάλωση ε, εκπομπή, ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να ε, σκεφτούμε μια συγκεκριμένη πολιτική για την Πολωνία. Είναι ίσως στη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη για την βιομηχανία που καταναλώνει η άνθρακα. Ευχαριστούμε ο Σφερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν ε, απορίες όπου οι περασπιστές ε, του συστήματος αυτού δεν μπορούν να απαντήσουν. Τι διευθυντικές αλλαγές ε, επετέφθησαν σήμερα με μέτρα ή καμία παρέμβαση στην αγορά. Τίποτα. Μηδέν. Ε, τι άνοιγμα υπάρχει στην προσέγγιση της αγοράς. Καμία. Μηδέν πάλι. Η αγορά ε, των δικαιωμάτων αυτών έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματικό και στρεβλό, διότι επιτρέπει αμύθιτα κέρδη σε κάποιους ε, καιροσκόπου και έχει πάρα πολλές αποτυχίες ελλείψεις και, και στήχησε και εκατοντάδε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους, στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, πρέπει λοιπόν κάτι να αλλάξει. Δεν μπορούμε να ε, συνεχίσουμε όπως ήταν τα πράγματα όπως προτείνουν οι πρασπιστές της αγοράς. Πρέπει να αλλάξει η προσέγγισή μας, να είναι ρυθμιστική και με κανόνε. Να είναι αποτελεσματική ω προ του περιβαλλοντικού ε, στόχου που θέλουμε να πετύχουμε και να είναι και δίκαιοι κοινωνικά. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος κύριος Κανιέτα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συζήτηση αυτή που έδειξε ότι έχουμε φτάσει σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό και τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Σημαντικός στάθμος ε, που έχει ήδη επιτευχθεί για τον ETS. Μπορούμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα και να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, σε μια πλήρη αρχιτεκτονική ε, του μηχανισμού ETS για την περίοδο μετά το 2020. Πέρυσι, εδώ μπροστά σας δεσμεύτηκα ότι τα στοιχεία του ETS, ό,τι αφορά το, ενεργεια... το πλαίσιο πλαίσιο για την ενέργεια να το ε, εξυγχρονίσω ε, από τη στιγμή που θα έχει εγκριθεί το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και δεσμεύομαι να το πράξω. Θα καταθέσω νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος ETS στις 15 Ιουλίου, άρα την επόμενη εβδομάδα. Μία πρόταση που θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ε, δουλειά μας για να πετύχουμε μια ενεργειακή ένωση και μια στραμμένη προς το μέλλον ενεργειακή πολιτική που είναι και προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούγκερ. Θα εστιάσουμε στις πτυχές των οποίων οι ευρωπαϊκοί μας έδωσαν σε καθοδήγηση τον Οκτώβριο του 2014. Πρώτα απ' όλα Έλε, δωρεάν κατανομή στο, ε, στη βιομηχανία. Αυτό θα συνεχιστεί ώστε εκεί που υπάρχει πραγματικά γνήσιος κίνδυνος διαρροής άνθρακα να ε, έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείες. Δεύτερον, εξυγχρονισμός, ταμείο εξυγχρονισμού για τον εξυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων για τα κράτη-μέλη με χαμηλότερο εισόδημα, δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εξυγχρονισμό τη παραγωγή ενέργεια σε αυτά τα κράτη-μέλη, είναι κάτι που επίση θα συνεχιστεί και η διαφάνεια έτσι θα βελτιωθεί σημαντικά. Τέλο, στήριξη για την ανάπτυξη καινοτομία για χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα θα συνεχιστεί μέσω του Ταμείου Καινοτομία ε, που θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή του και θα περιλάβει σχέδια καινοτομία για την βιομηχανία. Με αυτές τις προτάσεις μας πιστεύω ότι θα έχουμε μια ακόμη επικοδομητική πρόταση και συζήτηση. Θα συνεχιστεί ελπίζω και η συνεργασία που καθιερώσαμε εργαζόμενοι για αυτό το αποθεματικό και είμαι πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία για το κλίμα, για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και τους ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Ιβομπέλε, ηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σαφές ότι η πρόταση αυτή που θα ψηφίσουμε αύριο δεν είναι τέλεια, δεν θα μπορούσε να είναι τέλεια. Ξέρετε ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Είναι γνωστή αυτή η ρίση η καινοτομία, η χρηματοδότηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε βελτιώσει σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά πρόκειται για συμβιβασμό, όπω ξέρετε. Νομίζω ότι αξίζει να εγκριθεί από το σώμα αυτό ο συμβασμός, γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα μπρο ε, για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Η κυρία Γκέρλινγκ είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Όσοι επικρίνουν το σύστημα, έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, αλλά δεν προτείνουν καμία εναλλακτική λύση. Εντάξει, ωραία, μπορείτε να γκρινιάζετε, αλλά άμα δεν προτείνετε τίποτα άλλο, τι έννοια έχει. Δεν είναι επικοδομητική αυτή η στάση. Θα έλεγα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρήστε ότι κάναμε ό,τι μπορούμε. Δείξτε κάποια επίκαια, διότι στην Πολωνία και σε άλλα κράτη-μέλη ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές εξαιρέσεις και πρωτοβουλίες ε, μεταξύ αυτών των μέτρων, τόσο ώστε οι χώρες χαμηλού εισοδήματος να στηριχθούν τα κράτη-μέλη δηλαδή, όπου ο άνθρακας παίζει ακόμη πολύ σημαντικό ρόλο και η εξόριξή του. Και η Επιτροπή μόλις είπε ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις στον ενεργειακό τομέα ε, μέσω της αλληλεγγύης ε, που είναι σημαντικό ταμείο το Ταμείο Αλληλεγγύης για να βοηθήσει. Η επόμενη φάση λοιπόν θα είναι την επόμενη εβδομάδα 15 Ιουλίου θα κάνουμε μια δήλωση, θα υπάρξει μια δήλωση για τη μεταρρύθμιση του ETS, άρα δεν έχει τελειώσει αυτή την προσπάθεια. Όμως ε, κάνω έκκληση να μην είμαστε ιδιαίτερα αμυντικοί σε σχέση με αυτό, πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον και όπως είπε και ο Επίτροπος πρέπει να είμαστε επλεκτικοί. Πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις στους ενεργοβόρους κλάδους για να μην υπάρξει αυτή η περίφημη διαρροή άνθρακα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε γιατί είναι όντως ευάλωτοι. και εάν ε, δεν μπορέσουν να μεταφέρουν ε, το κόστος του ηλεκτρισμού τότε πρέπει να τους βοηθήσουμε. Φυσικά πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη, το καταλαβαίνουμε και μην ανησυχείτε, δεν είμαστε εχθροί του κλάδου. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Η συζήτηση για το θέμα αυτό ολοκληρώνεται. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη, που είναι η έκθεση Φερνάντες για τον προπολογισμό 2016. Εντολή για τον τριμερή διάλογο.